Okay, good afternoon everyone. I'm going to ask... Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε εδώ στην πρώτη σειρά, ώστε να μπορούν να σας δουν ε, όλους οι συνάδελφοί μας από τη Γάζα. Η αίθουσα είναι μεγαλύτερη από ό,τι σας δίνει η εικόνα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ σήμερα. Λυπούμαστε που δεν μπορέσατε να πάρετε βίζα για να έρθετε προσώπος, αλλά χαιρόμαστε που έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα αυτής της τηλεδιάσκεψης μαζί σας. Ελπίζουμε να διατηρηθεί το ρεύμα αρκετά, ώστε να μπορέσετε να συζητήσετε μαζί μας. Ε, εάν ε, όχι, ελπίζω να καταφέρουμε να ξαναέχουμε σύνδεση. Να σας ανακοινώσω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το υπόψη σας. Και για εκείνους από εσά που είστε εδώ θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον μπορείτε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε ενστάσει, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της προηγούμενης ε, συνεδρίασης. Σας έχουν διανεμηθεί, δεν υπάρχουν κάποιες ε, τροποποίησεις, επομένως θεωρούμε ότι εγκρίνονται και αυτά. Η διάσκεψη των Προέδρων έδωσε άδεια στην αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Παλαιστίνη για να ταξιδέψει το Φεβρουάριο του 2017 ε, σας ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ε, θα πρέπει να πούν στη γραμματεία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία. Υπάρχουν μόνο τέσσερις θέσεις διαθέσιμες, επομένως θα θέλαμε τουλάχιστον να υπάρχει εκπροσώπηση από τις πολιτικές ομάδες ή δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια συζήτηση για την κατάσταση στη Δυτική Οχθή και τις επικισμούς την τελευταία ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ε, ανακοινώθηκε και ψήφος επί του ζητήματος, αλλά δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα γίνει ψηφοφορία. Η ύπατη εκπρόσωπος κυρία Μοντεγκερίνη ήταν παρούσα για τη συζήτηση και ήταν παρούσα και για την προηγούμενη συζήτηση που είχε γίνει το Μάιο του 2016. Τα, ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου εξέφρασαν την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος ε, και δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση ή άλλη μορφή αντιστάθμισης από το Ισραήλ για την κατεδάφαση των ε, ε, έργων ε, που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο διάλογος έχει σταματήσει και συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε μορατόριο και εξακολουθούν να επεκτείνονται οι παράνομοι επικισμοί με εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους επίκους και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον στη Δυτική Όχθη. Ε, επηρεάζονται χιλιάδε Παλαιστίνοι από αυτές τι κατεδαφίσεις και τις υποχρεωτικέ μετακινήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ζητά να ξαναρχίσει η ειρηνευτική διαδικασία. Για την είπατε εκπρόσωπο, την κυρία Μεγερίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ο πιο συνεπής ε, χορηγός ε, στη διαδικασία της, ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής και τόνισε ότι ε, πρέπει να υπάρχει ενότητα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι κατά της ε, νομοθεσίας του Ισραήλ για τη ρύθμιση αυτή που υπάρχει για τις παράνομους επικισμούς ε, ε, στα παλαινιστινιακά εδάφη. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβουμε τα ενία, το επαναλάβαμε αυτό το Στρασβούργο και να βοηθήσουμε να υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία και για του Παλαιστινίου και για του Ισραηλινού. Συμφωνούμε ότι αυτό θα γίνει με τη συνεργασία των περιφερειακών εταίρων και οι Ηνωμένε Πολιτείε προφανώ και πρέπει να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά εμεί σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Κάνουμε έκκληση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να κάνει ό,τι της αναλλαγεί και θα θέλαμε να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν υπάρχει κάποια διαδικασία η οποία ε, έχει ξεκινήσει. Όσον αφορά την ε, δική μου την αποστολή στη Ραμάλα, στο συνέδριο της Φατάχ, είναι νωρίς ακόμα, ο, ο πρόεδρος Αμπάς ε, είναι ακόμα επικεφαλής ε, του ε, Φατάχ εγκρίθηκε ομόπονα από τα μέλη του συνεδρίου. Πολλά πράγματα με εντυπωσίασαν από αυτό το συνέδριο. Ένα ήταν ότι υπήρχε ειδικό τμήμα για τους 60 περίπου διεθνείς προσκεκλισμένους που προήλθαν από αρκετές χώρες, από την Κίνα, τη Βενεζουέλα, αρκετές αφρικανικές χώρες, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες. Ε, υπήρχε λοιπόν ε, διεθνή ελληνική η οποία προβλήθηκε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, στο συνέδριο αυτό καθεαυτό ήταν ότι η ηγεσία της Χαμάς έστειλε δήλωση στο συνέδριο και επίσης υπήρχε και εκπρόσωπος από εκπρόσωπους από άλλες ομάδες. Ε, υπάρχει μια διαδικασία συμφιλίωσης, υπάρχει διεθνής αλληλεγγύη από τις αντιπροσωπείες, από τους ευρωβουλευτές τες που ήταν εκεί παρόντες και φυσικά και εγώ εξέφρασα ε, και ε, την αλληλεγγύη μας εξ ονόματος όλους και εξ ονόματος ε, της δικής μου της πολιτικής ομάδος. Υπάρχει υποστήριξη λοιπόν η οποία έτυχε θερμής υποδοχής. Υπάρχουν δύο αμφιλεγόμενες ψηφοφορίες, ε, ε, το ε, ψήφισμα για το θόρυβο και το ψήφισμα για τη ρύθμιση των παράνομων επικισμών. Ε, αναμένεται να γίνεται σήμερα αρχική ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν υπάρχει επικέρωση, ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη. θα δούμε τι ακριβώς συνέβη και υπάρχουν και εκκλήσεις... Ε, για, ε, από την πρωινή προσευχή για να σταματήσουν τα ηχεία ε, πρόταση προς τους Παλαιστινίους που λέει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και εγώ συμφωνώ βέβαια από αυτού. Οι επικισμοί και οι κατεδαφίσεις αναμένεται να συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Στην πρώτη ανάγνωση του ε, νομοσχεδίου για την νομοποίηση 4.000 αυθέρωτων ε, κατοικιών στη Δυτική Όχθη. Εδώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ομόφωνα κατά αυτού του νομοσχεδίου και ε, καταδικάζει την υποκλοπή αυτή της ιδιωτικής γης και υπάρχουν και φόβοι ότι θα ξεκινήσει και έρευνα και ότι ε, ο Ομπάμα θα αναλάβει δράση. Ε, υπάρχουν κάποιες διαρροές στον τύπο ε, και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και την αντίθεση που υπάρχει για αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει ο Δήμος της Ιερουσαλήμ, ο οποίος έχει περίπου ε, παράνομους επικισμούς στο 75% ιδιωτικών κατοικιών Παλαιστινίων. Η Πισνάου, μη κυβερνητική οργάνωση, είπε ότι η νομοθεσία αυτή στην ουσία θα νομιμοποιήσει 55 επικισμούς, 4.000 επίκους παράνομος φυσικά. Η Peace Now λέει ότι πρόκειται για αρπαγή για κλοπή και επίσης κλέβει και αποστερεί και από τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους την δυνατότητα να καταλήξουν σε μία λύση ανάμεσα σε δύο κράτη. Το ίδιο και ο Δήμος της Ιερουσαλήμ έχει ανανεώσει το σχέδιό του για την ε, κατασκευή άλλων 500 κατοικιών στο Ραμάτ Σλόμο. Ταυτόχρονα υπήρξαν και πάρα πολλές κατεδαφίσεις το 2016, προσπαθούν να ελέγξουν τις στρατηγικές θέσεις, ε, τις στρατηγικές θέσεις για να ευνοήσουν τους επίκους. Νέες 770 κατοικίες επίσης θα οικοδομηθούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όπως είπα, οι 500 έχουν ήδη προχωρήσει στο Ραματσλόμο. Πάντα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά βέβαια αντιμετωπίζουν την κριτική της διεθνούς κοινότητας γιατί επηρεάζει την ιδιοκτησία της γης στην περιοχή και αλλοιώνει την πληθυσμιακή σύνθεση. Είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την συνέχεια μιας μελλοντικής, την εδαφική συνέχεια, μιας μελλοντικής παλαιστινιακής κρατικής οντότητας. Τώρα βέβαια αυτή η δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και πάρα πολύ έντονη Πάντως ε, λέγουν ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε δράση για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο ε, κρατών. Πού είναι δυστυχώς η πολιτική βούληση που θα επέτρεπε να επηρεάσουμε τα πράγματα όπως το ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει ας προχωρήσουμε τώρα ε, για να δούμε την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση στη Γάζα θα προσπαθήσουμε επίσης στην επόμενη αποστολή μας όταν πάμε τον Φεβρουάριο στην Παλαιστίνη να ξαναπάμε στη Γάζα. Κάθε προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα απερίφθη. Όπως γνωρίζουν τα μέλη ε, δεν μας δόθηκε άδεια εισόδου και διαμονητήρια στην Γάζα. Ήδη από το 2011 τρέχει αυτή η ιστορία. Υπήρξε μια πάρα πολύ σύντομη επιτόπου επίσκεψη από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον κύριο Ζων Αρτουή. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό μαζί του. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους προσεκλημένους μας για να δούμε ποια είναι πραγματικά η ζωή στη Γάζα σήμερα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές που έχουμε μπροστά μας, στον Γκάιλ Λέοπολντ που είναι υπεύθυνο ε, της Premier Urgence Internationale για την Παλαιστίνη. Χαίρομαι που σας βλέπω. Επίσης έχουμε και τέσσερις ομιλητές από τη Γάζα. Καταρχάς ο συντονιστής της Premier Urgence Internationale, Έχουμε ένα γεωργό, έχουμε μία γυναίκα η οποία ασχολείται με την αλληλεία. Um, what we're going to do, I going... Και έχουμε και την Πατρίσια Γκρίλο. Θα ξεκινήσω λοιπόν, συγγνώμη μια στιγμή γιατί έχω λίγο μπλέξει τους καταλόγους μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν Ο Μοχάμεντ Αλμπάκη, Μοχάμεντ Ελμπάκρη μάλλον, διαχειριστής των Επιτροπών Γεωργίας. Σας καλωσορίζω όλους στην συνάντηση αυτή. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον πληθυσμό ε, της Γάζα ε, που φτάνει τα 2 εκατομμύρια, έφτασε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε για τη γέννηση ενός αγοριού. Δυστυχώς ο αποκλισμός της Γάζα έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη της Λωρίδας. Έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια τρεις εισβολές πολεμικές και αυτό έχει πάει πολύ πίσω τα πράγματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανεργία στη Γάζα είναι 42%. Το 80% των κατοίκων της Γάζα παίρνουν κάποια βοηθήματα. Η φτώχεια είναι πάρα πολύ υψηλή και το 90% των κατοίκων της Γάζα δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Συναντηθήκαμε και με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος για τις συνέπειες που έχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην υγεία των ανθρώπων και τη ζωή τους. Έχουμε 65.000 εκτοπισμένους και θέλουν βοήθεια για να ξαναχτίσουν τα κατεστριμμένα σπίτια τους. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η κατάσταση στη Γάζα είναι μια ορολογιακή βόμβα. Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα πώς είναι η ζωή μέσα στη Γάζα και τι μπορούμε εμείς ε, για να βοηθήσουμε. σαν κοινοβούλιο, σαν επιτροπή κτλ. Θέλετε εσείς να αποφασίσετε το ποιος θα ξεκινήσει ή να δώσω Κοιτάξτε, ο Γκαέλ θα πάρει το λόγο και μετά η Πατρίσια και μετά θα μιλήσετε εσείς. Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι, σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζα. Όπως η Urgency International την διαπιστώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ευχαριστήσω την κυρία Άντερσον, την κυρία Ζάμιτ και τον κύριο Λαυσνιούσεν και την επιμελητία και διερμηνία και εδώ και στη Γάζα που καθιστούν τη συνάντηση αυτή εφικτή. Το ότι είμαστε εδώ σήμερα είναι κάτι που με θλίβει. Με θλίβει γιατί η παρουσία μας εδώ είναι συνέπεια της αδυναμίας μας να πάρουμε τις θεωρήσεις έτσι ώστε οι συνάδελφοι από τη Γάζα να έρθουν εδώ σήμερα. Για να φύγουν από τη Γάζα και να έρθουν εδώ, ένας κάτοικος πρέπει να αποκτήσει μια Ισραηλινή άδεια για να πάει στα σύνορα με την Ιορδανία. Πρέπει να έχει μια επιστολή των Ιορδανών ότι συμφωνούν για την είσοδο στην Ιορδανία και μια βίζα Σέγγεν. Από τα τρία αυτά έγγραφα και παρά τη βοήθειά σας και τη βοήθεια του γαλλικού προξενείου πήραμε μόνο τη βίζα. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, γιατί ακόμα και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη είδαν ότι το ποσοστό άρνησης των δικών τους αιτήσεων από 3 πήγε σε 21% το 16%. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση η οποία δείχνει την φρικτή καθημερινότητα την οποία αντιμετωπίζουν οι Γκαζαούοι που υφίστανται τον αποκλεισμό των Ισραηλινών εδώ και 10 χρόνια. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιους αριθμούς από τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Η Γάζα σήμερα τι είναι. Ένας ε, αποκλεισμός σε ένα έδαφος 40 ε, χιλιόμετρων μήκους και 15 ε, χιλιόμετρων πλάτους με 2 εκατομμύρια κατοίκους. 80% των κατοίκων που ζουν με βοηθήματα και ιδιαίτερα με τρόφιμα. 46% έχει αβεβαιότητα για την έβρεση τροφίμων. Το ποσοστό ανεργίας είναι 42% και στους νέους φτάνει το 60%. 75% ε, του πληθυσμού αντιμετωπίζει φρικτά προβλήματα υγείας λόγω του βρώμικου ύδατος. Το 60% του νερού που καταναλώνεται δεν είναι πραγματικά πόσιμο. Ε, πραγματικά επίσης ε, χύνονται στη θάλασσα 36 Ολυμπιακές πισίνες απόβλητα την ημέρα. 6 με 10 ώρες την ημέρα ηλεκτρικό. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή των Καζαουή αλλά και την οικονομία της περιοχής. 70.000 ζουν σε προσωρινές κατοικίες γιατί έχασαν τα σπίτια τους στη σύγκρουση του 2014. Τους ε, είχαν υποσχεθεί το 2014 στο Κάιρο ε, πολλά χρήματα, αλλά έχουν πάρει μόνο το 40% μέχρι πριν από λίγους μήνες. Μία λίστα απαιτήσεων από πλευράς του Ισραήλ για εισαγωγή προϊόντων, απαγορεύεται η εισαγωγή νερού, τροφίμων, πολλές φορές ε, εμείς δεν μπορέσαμε να στείλουμε σαν παράδειγμα αντλίες για να τραβήξουν νερό από ε, μεγάλη απόσταση σε βάθος. Νομίζω ότι υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά προβλήματα περιορισμού κίνησης και των αλλιέων. Δεν μπορούν παρά να χρησιμοποιήσουν οι αλλιείς παρά μόνο το 15% των αλλιευμάτων που τους ανήκουν. Το 2020, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, η περιοχή δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμη και η Παγκόσμια Τράπεζα μιλάει ήδη για έκρηξη στην περιοχή και ο ΙΕ μιλάει για ορολογιακή βόμβα. Η κατάσταση στη Γάζα βέβαια δεν είναι τόσο άσχημη όσο στη Συρία και το Ιράκ. Μην ξεχνάμε όμως ότι ένα παιδί στη Γάζα 10 ετών σήμερα έχει ζήσει τρεις πολέμους με το Ισραήλ, ένα αιματηρό εμφύλιο και 15 χρόνια εμπορικό αποκλεισμό και ναυτικό αποκλεισμό επίσης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την μαζική ε, αφήξη ε, μεταναστών και δεν υπάρχουν κάτοικοι από τη Γάζα βέβαια γιατί το Ισραήλ ελέγχει και αποκλείει την περιοχή της Λωρίδας. Αυτό πραγματικά δεν προμηνύει τίποτα καλό για τη Γάζα, τους κατοίκους της και την περιοχή. Μόνο αν αρθεί ο εμπορικός αποκλεισμός και η πολιτική λύση θα επιτρέψουν να μην συνεχιστεί η χειροτέρευση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης, κυρίως όμως της ανθρωπιστικής κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε. Ε, ζωφερά, το λιγότερο που μπορώ να πω αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές και να πηγαίνουν και προς τα έξω. Θα δώσω το λόγο στο Τζιχάντα Μπιχάσεν, ο οποίος ε, είναι ο ε, υπεύθυνος συντονισμού στη Γάζα, για να ε, μιλήσει για περίπου πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ζιχάδα Μπιχάσαν, είμαι ο συντονιστής επιτόπου εδώ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έρθουμε να σας δούμε εκεί για να σας περιγράψουμε την πραγματικότητα στη Γάζα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα σας μιλήσω Συντεμία, για την παρέμβασή μας ε, για την ε, περιοχή αυτή στην οποία υπάρχει πρόσβαση. Είναι μια περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, περίπου 300 μέτρων, στην ανατολική πλευρά της Γάζας, από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι μια περιοχή στην οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχει ένας φράχτης ε, και περίπου 1500 μέτρα από το φράχτη υπάρχει κίνδυνος για τους ε, πολίτες. Μετά από το 2008 το Ισραήλ περιόρισε την πρόσβαση από τα 300 μέτρα στα 100 μέτρα μόνο για τους γεωργούς. αλλά οι γεωργοί στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν πάντα απειλές όταν ε, προσπαθούν ε, να πάνε στα χωράφια τους. Οι Ισραηλινοί επικαλούνται λόγους ασφαλείας και χρησιμοποιούν ε, πραγματικές σφαίρες και πυροφολούν σε αρρώσιμες εκτάσεις ε, τις οποίες καλλιεργούν αυτοί οι γεωργοί. Ε, χρησιμοποιούνται επίσης ψεκασμοί επικίνδυνων ουσιών στις ε, ε, εκτάσεις αυτές, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και γενικώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση οι γεωργοί στη γη τους. Από τις αρχές του 2016 είχαμε 20 τραυματισμούς ε, αλλιέων και 5 γεωργών. Οι γεωργοί καλλιεργούσαν σε αυτά τα 300 μέτρα ε, και γενικότερα βρίσκονται ε, σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από το φράχτη. Οι γεωργοί λοιπόν σε αυτή την περιοχή, την περιορισμένη ζώνη, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες, μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. έχουν μεγάλους περιορισμούς και δυσκολεύονται πολύ ε, να φτάσουν ε, στη γη τους. Εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμα και σήμερα και πιστεύουμε πραγματικά ότι η κατάσταση στη Γάζα ε, όσο αυξάνεται η υποτιθέμενη προστασία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και αυτό φυσικά ε, έχει σχέση με, τους, ε, με το καθεστώς κατοχής και την κατάσταση στη Γάζα. Εάν δεν σταματήσει λοιπόν πλήρως ε, αυτός ο αποκλεισμός, η Πρόεδρος, μήπως θα μπορούσαμε να ακούσουμε Μία από τις δύο κυρίες που έχουμε εδώ μαζί μας, ε, την κυρία Μπουτία Ρίσος, η οποία είναι γεωργός. Θα σας ευχαριστώ. Είμαι γεωργός. Το σπίτι μου βρίσκεται στα 800 μέτρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Δεν είναι της ιδιοκτησίας μου, ενοικιάζω αυτή τη γη και το αγρόκτημά μου βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το φράχτη που βρίσκεται στα σύνορα. Είμαι εκεί με το σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Δυσκολεύομαι να βγω και από το σπίτι μου, τα παιδιά μου επίσης και θα ήθελα Η πρόεδρος διακόπτη μπορείτε να μιλείτε λίγο πιο αργά για να μπορούν να σας προλαβαίνουν ε, οι διερμηνείς. Να πλησιάσετε λίγο πιο καλά στο μικρόφωνο και να μιλάτε λίγο πιο αργά. Είμαι γεωργός εδώ και 16 χρόνια. Ανέθρεψα τα παιδιά μου, τα έστειλα στο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά χάρη στη δουλειά μου, από τη γη, ε, από τη γη που καλλιεργώ. Όλοι οι πόλεμοι, οι εισβολές, αυτό το καθεστώς κατοχής ε, μας βομβάρδισαν, μας χτύπησαν και με πυράβλους ε, στα 8, στα 12 μέτρα και όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν και τη γη και εμείς την νοικιάζουμε αυτή τη γη το έδαφος ε, δεν είναι πλέον ε, γόνιμο για να καλλιεργήσουμε και δεν ε, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τόσο εύκολα. Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Είτε το δίκτυο ίδρευσης, τα αρτεσιανά πηγάδια, οτιδήποτε έχουμε, όλα αυτά έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς. Και όταν δεν υπάρχει έφορο έδαφος για να καλλιεργήσουμε, Μπορεί να φταίει ορισμένες φορές η φύση, αλλά φταίει και η ποιότητα του νερού, έχουμε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, έχουμε συνεχώς ε, διακοπές ρεύματος. και το δίκτυο ίδρυυσης ε, ορισμένες φορές παρέχει πάρα πολύ ζεστό νερό, νερό το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις καλλιέργειές μας. Σας μιλώ με κάθε ειλικρίνεια. Ζούμε πάρα πολύ δύσκολα, απλώς ο χρόνος κυλάει. Μέσα σε ένα μήνα έγιναν διάφορες επιθέσεις από αέρος, με διάφορα αεροσκάφη και ψεκασμοί. Και αυτό φυσικά επηρεάζει και τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, χρειαζόμαστε φυτοφάρμακα. Τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά, στοιχίζουν 400 δολάρια, 500 δολάρια. Και δυστυχώς ε, δύσκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ε, ε, έχω τεράστια χρέη και δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε καν να πουλήσουμε τα προϊόντα μας ε, πάρα πολύ ακριβά. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Ζούμε σε ένα καθεστώς μόνιμου φόβου και πανικού. Θέλουμε απλώς να ζήσουμε με ασφάλεια και ειρήνη. Αλλά δεν μπορούμε καν να ανάψουμε φως ε, στην αυλή μας, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η περιοχή αυτή ήταν γεμάτη αγροκτήματα, μπορούσαμε να πουλήσουμε και τα προϊόντα μας ε, με σχετική ευκολία, αλλά από το Μάιο και μετά αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες και τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Αντιμετωπίζουμε πάσης φύσεως δυσκολίες. Χάσαμε ε, ε, εκτάσεις, 12 ε, στρέμματα εγώ, τρακτέρ, υπάρχουν ε, οι φράχτες, υπάρχουν σημεία ελέγχου. Είναι αδύνατον πλέον να εργαστούμε. Το 2008 τα παιδιά μου ήταν μικρά. και τότε αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες, ε, μπήκαν οι στρατιώτες μέσα στο σπίτι μας ε, δια της βίας και ακόμα και τώρα που ενηλικιώθηκε η κόρη μου ε, κάθε φορά που ακούει θορύβους από το σοκ τότε κρύβεται. Ένα από τα παιδιά μου έχει καταντήσει επέτησα και συγγνώμη, δεν μπορεί, έχει τραυλίζει δεν μπορεί να μιλήσει από το σοκ. Παρόλα αυτά εμείς προσπαθούμε ακόμα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να συνεχίσουμε ε, τη ζωή μας. Τίποτα άλλο. Could, uh, could η Μαντλίν να μιλήσει για τη δική της δραστηριότητα. Είστε η μόνη γυναίκα που ασχολείται με την αλληλεία στη Γάζα. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας εμπειρίες. أول سيارة طبعا فلسطين Έχουμε προβλήματα όπως ακούσατε στη γεωργική παραγωγή στην Γάζα αλλά έχουμε προβλήματα και στην Αλία. Δεν είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε τα ύδατα τα οποία μας ανήκουν. Εμείς προσπαθούμε να πάμε σε περιοχές όπου υπάρχουν πλούσια αλλιεύματα. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε εδώ και δεκαετίες, αλλά δυστυχώς σε αυτές τις ζώνες οι Ισραηλινοί έχουν αποκλείσει την πρόσβασή μας. Είναι αδύνατο για τους αλληλείς να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν. για τις Σαρδέλες ας πούμε θα πρέπει να φτάσουμε στα 6 μίλια από την ακτή, αλλά δυστυχώς οι Ισραηλινοί δεν μας αφήνουν να ξεπεράσουμε τα 5. Όταν λοιπόν εμείς σαν αλληλείς ε, βγαίνουμε με τις βάρκες μας, δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, δεν ξέρουμε καν αν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε τα σκάφη μας με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουμε είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, δεν μπορούμε να τα ανακαινήσουμε και ένα μεγάλο ποσοστό των αλλιέων λόγω του εμπορικού αποκλεισμού δεν είναι καν σε θέση να εξάγουν τα αλλιεύματά τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών μας υποχρεώνουν να μένουμε στα δύο μίλια από την ακτή, ακόμα χειρότερα δηλαδή από ό,τι παλιά. Κάτι το οποίο καθιστά τη δραστηριότητά μας εξαιρετικά δύσκολη. Και δυστυχώς έχουμε και πάρα πολλούς αλληλείς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μας χτυπάει η αεροπορία του Ισραήλ. Πολλές φορές υπάρχουν ε, διάφοροι σκοπευτές τη στιγμή που πλησιάζουμε στην ακτή. Και γνωστοί μου έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας φίλος μας μάλιστα δεν μπόρεσε να επιστρέψει ε, στον σωστό χρόνο, στη σωστή τοποθεσία, όπως ήταν υποχρεωμένος και αυτό οδήγησε στο να χάσει τη ζωή του δυστυχώς. Και υπάρχουν και πάρα πολλά ατυχήματα στην αποκλεισμένη περιοχή από τους Ισραηλινούς και από τα ηλεκτροφόρα σύρματα, καταλήγουμε στο νοσοκομείο και όπως είπα δεν είμαστε προστατευμένοι και από αδέσποτα πυρά. Εμένα προσωπικά μου έκλεψαν, μου κατέσχεσαν την βάρκα μου, μου κατέσχεσαν τα δίχτυα που είχα πάνω στη βάρκα, μου τα έκλεψαν ουσιαστικά. Και οι Ισραηλινοί μας κατηγορούν ότι πηγαίνουμε και ψαρεύουμε ακριβώς στα όρια. Μα τι άλλο να κάνουμε, πού αλλού να πάμε για να ψαρέψουμε. Όπου και να είμαστε, στα όρια είμαστε. Είτε προς το νότο είτε προς το βορρά, τα όρια δυστυχώς είναι πάρα πολύ στενά για μας. Άλλωστε πολλές φορές που ψαρεύω αρκετά μακριά από τα σύνορα τα λεγόμενα, δυστυχώς ανάλογα με τον καιρό ε, μπορεί να μετακινηθούμε χωρίς να ελέγχουμε απόλυτα την τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε. Όλα αυτά κάνουν τη δραστηριότητά μας επισφαλή και κουραστική. Όπως είπα, χάνουμε συχνά τα πλοία μας, τα οποία τα κατάσχουν οι Ισραηλινοί και επίσης και τα δίχτυα. Και χρειάζονται πέντε χρόνια για να το ξαναπάρουμε πίσω. Και όταν καταφέρνει κάποιος ε, ψαράς από τη Γάζα να πάρει πίσω το σκάφος του, ε, είναι σε κακοχάλι, τίποτα δεν δουλεύει. Θυμίζω ότι είναι συνθετικές κατασκευές αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούμε πια, εξαιρετικά κακής ποιότητας, δεν είμαστε σε θέση να τα συντηρήσουμε, δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε τίποτα που να μας βοηθήσει εν βάση περιπτώσει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Και δεν μας επιτρέπουν να βρούμε τα ανταλλακτικά που μας είναι απαραίτητα. Και η μεγάλη ταλαιπωρία είναι τα δίχτυα. Εγώ έχω δίχτυα πέντε χρόνια τουλάχιστον τα ίδια και δεν καταφέρνω να τα αλλάξω γιατί δεν μπορώ να τα βρω, δεν υπάρχουν, δεν εισάγονται. Συνεπώς λοιπόν η δουλειά μου η οποία κανονικά θα έπρεπε να ζει την οικογένειά μου αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε ένα συνεταιρισμό και ο συνεταιρισμός με βοήθησε και έτσι κάπως επιβιώνουμε οικονομικά εγώ και η οικογένειά μου. Η τράπεζα, η κεντρική τράπεζα της Παλαιστίνης μου έδωσε ένα δάνειο 4.000 δολαρίων και ελπίζω να μπορέσω να επισκευάσω το σκάφος μου και να μπορέσω να ξαναρχίσω την αλληλεία γιατί όπως σας είπα δεν είχα αυτή τη δυνατότητα τους τελευταίους μήνες. Όλα είναι ακριβά και δύσκολα για μας. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε δυστυχώς όσο και αν ακούγεται περίεργο είναι πανάκριβα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα ζητήσω από την Πατρίσα Γκερίλο να μιλήσει για πέντε λεπτά και μετά θα ξαναδώσουμε και πάρει το λόγο. Ο Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ήρθε, ε, η Αντιπρόεδρος και θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για κάποιες ερωτήσεις. Κυρίες και κύριοι, το ερώτημα πλέον είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Στις διάφορες παρεμβάσεις το ακούσαμε. Το 70% των κατοίκων της Γάζας εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο αποκλισμός, ε, η κατάρρευση της οικονομίας ε, δεν επιτρέπει καμία εξέλιξη και οικονομική ανάκαμψη και έχει φυσικά καταστροφικές ε, ανθρωπιστικές συνέπειες. Πιστεύουμε ως άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε επιτόπου, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να συμβαδίζει με πολιτικές δράσεις για πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Η Γάζα είναι απόσπαστο τμήμα των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά από τη Δυτική Όχθη μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις ε, και αυτές τις πολύ ισχυρές μαρτυρίες ε, της ε, Ματλίν και της Βέζενταν, θα επικεντρωθούμε σε τρεις κυρίως τομείς. Στον αποκλεισμό, στους, στις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ο αποκλεισμός θα είναι δεκαετής πλέον του χρόνου. Θέλετε πραγματικά να περάσει άλλη μια δεκαετία αποκλεισμού. Η απάντηση φυσικά είναι αρνητική. Γι' αυτό και ακριβώς ε, σας προτρέπουμε να μην ε, ε, ξεχάσετε τη Γάζα και να δράσετε το Ισραήλ ε, κάνει πράγματα τα οποία ε, καταδικάζονται από το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει ο αποκλεισμό για να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις και να διευκολύνει το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτών των ανθρώπων και αγαθών επίσης από και πριν ε, και προς τη λωρίδα της Γάζας. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσει για μια βιώσιμη οικονομία. Ο αποκλεισμός αυξάνει την ε, επισητιστική ανασφάλεια και επίσης υπονομεύει την πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια και σε υπηρεσίες παιδείας. Ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν με συγκεκριμένο στόχο να σταματήσει αυτός ο αποκλεισμός ανανεώνοντας τις πιέσεις προ την Ισραηλινή κυβέρνηση, να σταματήσει την πολιτική της και να αλλάξει πολιτική ενώπιον της Γάζας. Ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ε, της υπάτης εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής ασφαλείας ε, στις συζητήσεις για την ε, ειρηνευτική διαδικασία την οποία ξεκίνησε η Γαλλία και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα θα βρίσκεται ε, μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων. Όσον αφορά την ε, περιοχή αυτή της περιορισμένης πρόσβασης, ε, σας το παρουσίασε η Βεζεντάν και η Ματλίν και ο Τζεχάντ. Η πρόεδρος ρώτησε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή, η οποία τιμωρείται διπλά. Από τη μια υπάρχει ο και από την άλλη υπάρχουν και άλλοι περαιτέρω περιορισμοί το γεγονός ότι οι γεωργοί και αλληλείς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γη τους και να έχουν πρόσβαση σε ελευτικές ζώνες παραβιάζει αρκετές διατάξεις διεθνούς δικαίου. Η εφαρμογή της ζώνης Α ε, έχει αφήσει τις γεωργικές αυτές κοινότητες σε κατάσταση φρικτής φτώχειας. Επιπλέον, το θέμα της προστασίας των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό ήταν σαφέστατα από τις μαρ... σαφέστατο από τις μαρτυρίες που μόλις ακούσαμε. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται αληθινά πυρά ε, και χημικοί ψεκασμοί για τις καλλιέργειες ε, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη δουλειά των ανθρώπων που ζουν εκεί. Ζητάμε λοιπόν από το Κοινοβούλιο να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν, να πιέσουν την Ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε πρώτον να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση και ελεύθερη κυκλοφορία για τους ανθρώπους που εργάζονται και ζουν εκεί και δεύτερον να σταματήσουν να πυροβολούν ε, γεωργούς, αλληλείς, πολίτες εν γέννη. Τέλος, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ε, κρίση λογοδοσίας που υπάρχει στα ε, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στη λωρίδα της Γάζας. Ε, ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να προστατεύει τους Παλαιστινίους πολίτες και επίσης όλες οι χώρες έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύνεπώς, ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να πιέσουν την Ισραηλινή κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της η συνεχής επιδείνωση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας και της ζωής δύο εκατομμυρίων ανθρώπων ε, δεν είναι αποδεκτή. Η Γάζα και οι άνθρωποι της δεν θα μπορέσουν να αντέξουν άλλη μία δεκαετία αποκλεισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εντάξει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, για αυτές τις πολύ σημαντικές συνεισφορές και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους υπολείπους γιατί ό,τι είπε η Πατρίτσια και ό,τι ακούσατε προηγουμένως με βρίσκουν σύμφωνοι. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω ε, για τις εκκλήσεις που κάνετε προς το Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους Ευρωβουλευτές ε, και στους υπολείπους. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις όλων. Να χαιρετήσω αδελφικά τους φίλους από τη Λωρίδα της Γάζα. Να πω ότι δεν μπορούμε πια, όλα τα ίδια ακούμε. Ζητάμε από διάφορες αρχές και υπηρεσίες στον κόσμο με τη Μαρτίνα είχαμε πάει πέρυσι στο Ισραήλ, θελήσαμε για μια ακόμη φορά να πάμε στη Λωρίδα. Μα ε, μας απαγόρευσαν φυσικά να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να σας περιγράψω τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και τις οποίες μας δημιουργεί το κράτος του Ισραήλ. Νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πάψουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να σταματήσουν τη σιωπή τους, γιατί η σιωπή τους πια κρατάει πολύ καιρό και έχει αρχίσει και γίνεται εκοφαντική. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Μαρτίνα. Να στείλουμε μια επιστολή επίσημη στους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων έτσι ώστε επιτέλους να απελευθερωθεί η Γάζα και να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί να ζήσουν εν πάση περιπτώσει. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα δούμε από τις αντιδράσεις τους. Το να το κάνουμε αυτό, τη συζήτηση αυτή και να ζητάμε μόνο από τις Βρυξέλλες να αντιδράσουν δεν αρκεί. Λοιπόν, είναι μια ιδέα την οποία άκουσα και τη μεταφέρω γιατί πρέπει και εμείς να την εφαρμόσουμε. Έχετε το λόγο απέναντι. Ναι, είμαι ο Σωτήρος Δαγιανόπουλος, ε, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Παίρνω το λόγο γιατί ε, πριν μερικές μόλις μέρες ήμουν και εγώ στην Ραμάλα της Παλαιστίνης μαζί με την πρόεδρο εδώ της αντιπροσωπείας τη Μαρτίνα την Άντερσον στο συνέδριο της Αλφατάχ. Και πριν πάω στις ερωτήσεις και προς τους φίλους και φίλες από την Παλαιστίνη να πω δύο πράγματα σαν εντύπωση. Για πολλωστή φορά γιατί και πέρσι ήμουν εκεί και άλλες φορές. Είναι πραγματικά ε, συγκινητικό και μεγάλο δίδαγμα και για τους ευρωπαϊκούς λαούς ένας λαός όπως ο Παλαιστινιακός που 100 χρόνια τώρα τον σφάζουν θα θυμίζω ότι ε, το 1917 ξεκίνησε το κυνηγητό των Παλαιστινίων με την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ, συνεχίζει να έχει ακόμα τόσο μεγάλη πίστη και τόσο μεγάλο ενθουσιασμό για την νίκη του. Δεύτερη παρατήρηση, ότι πραγματικά πρέπει να το ζήσεις και να το δεις από κοντά την κατάσταση που υπάρχει εκεί και που δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν έχεις ιδιωτελή συμφέροντα και πολιτικά συμφέροντα να μην αναγνωρίζεις ότι πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταστάσεις στον κόσμο. Είναι κατοχή, είναι apartheid, είναι μεθοδευμένη εδώ και πολλά χρόνια προσπάθεια να εξαφανιστούν οι Παλαιστίνοι από τη γη τους. Ή να μεταβληθούν όλοι σε πρόσφυγες, όπως τόσοι πολλοί μέχρι τώρα, ή κυριολεκτικά να γίνει γενοκτονία. Πάω λοιπόν στις ε, ερωτήσεις πολλές φορές και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου και των κυβερνήσεων και σε συναντήσεις στην, στην Παλαιστίνη δηλώνεται η βούληση πολλών κυβερνήσεων ε, να σταματήσει ο αποκλεισμό, να σταματήσουν οι επικισμοί, να σταματήσει η κατοχή και όλα αυτά. Και μάλιστα δηλώνεται και η βούληση να αναγνωριστεί από τις κυβερνήσεις το Παλαιστινιακό κράτος που ξέρετε ότι ελάχιστα κράτη το έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα. Ελάχιστα όλα αυτά, τίποτα πολίτε δεν προχωράει από όλα αυτά. Μένουν μόνο στα λόγια. Και βεβαίω αυτό το γεγονό ενισχύει την επιθετικότητα του Ισραήλ. Ακόμα περισσότερο. Οι πιέσει, όπω λέγονται, των κυβερνήσεων ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλήγουν απολύτω πουθενά γιατί οι κυβερνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να καταλήξουν πουθενά και έρχομαι στην ερώτηση που αφορά και του συναδέλφου μέλη του Ευρωκοινοβουλίου αλλά κυρίω του φίλου και του φίλες που μα ακούνε, ελπίζω να μα ακούνε στην, ε, στη Γάζα. Η ερώτηση είναι η εξή. Μετά από όλε αυτέ τι δηλώσει κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών οργάνων που δηλώνουν αλληλεγγύη ε, και πρόθεση αναγνώριση του κράτους της Ισραήλ κτλ. Αν αύριο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δηλώνουν αυτή την πρόθεση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση που δηλώνει αυτή υποτίθεται την πρόθεση αν αύριο διέκοπταν όλων των ειδών τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Εμπορικές, διεθνείς, οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτικές. Πόσο καιρό θα έπαιρνε με τέτοια σοβαρή πίεση στο κράτος του Ισραήλ για να γίνει ένα βήμα στην λύση του προβλήματος. Θα ήταν ένα χτύπημα σε αυτή την πολιτική του Ισραήλ και μια βοήθεια, πραγματική βοήθεια στους Παλαιστινίους και θα έδινε φτερά στον αγώνα τους. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και θα ήθελα και τη γνώμη των ε, φίλο μας από την ε, Γάζα. Ε, Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω μία πρόταση απευθείας. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους προσκεκλημένους μας. Τους εύχομαι να αντέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Εμείς Είμαστε δίπλα τους. Και ως πρόταση θα ήθελα να ζητήσω από την αντιπροσωπεία να γράψουμε στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, στην Κνεσέτ, και να ζητήσουμε σε όσους από τους Ισραηλινούς βουλευτές θελήσουν να έρθουν, ε, να έρθουν για να μας μιλήσουν για αυτό το νόμο, ο οποίος θα έχει και αναδρομική ισχύ για τους επικισμούς ε, και φυσικά ε, θα έχει σοβαρές ε, και οικονομικές συνέπειες. Ε, να πιέσουμε δηλαδή και από πλευράς μας το Ισραηλινό Κοινοβούλιο ώστε να σταματήσει ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου. Ναι, χαίρετε. Εγώ ήρθα πριν από 10 λεπτά και έτσι έχασα κάποια από τα πράγματα τα οποία συζητήσατε αλλά ήταν ε, ενδιαφέρον, όπως είπε και κάποιος ε, κάποια στιγμή εδώ, ότι εμείς εδώ, σε αυτή την αντιπροσωπεία, πραγματικά στικόμαστε δίπλα σας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας, αλλά πρέπει να είμαστε μια ευρύτερη δύναμη ισχύω εάν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Εγώ είμαι Σουηδή σοσιαλδημοκράτη. και όπως ξέρετε η Σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε όταν ε, αναλάβαμε την εξουσία πριν από ένα-δύο χρόνια να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Θα μπορούσαμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι υπάρχει ε, μια σειρά πολύ ισχυρών ψηφισμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στα οποία έχουν ψηφίσει πάνω από 500 βουλευτές υπέρ μιας στεναρής θέσης. Ανέκαθεν λοιπόν προσπαθούσαμε να βρούμε και προσπαθούμε ακόμα ε, να βρούμε περισσότερα μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε θεσμικά όργανα εκτός του Κοινοβουλίου αλλά ε, και γενικώ ε, φορείς τους οποίους μπορούμε να βασιστούμε που μπορούν να δώσουν και σε εμά και σε εσά μεγαλύτερη αξιοπιστία και δύναμη ισχύω. Βεβαίως και θα μιλήσω με την Σουηδή Υπουργό Εξωτερικών, μια γυναίκα η οποία ήταν ε, αυτή η οποία υποκίνησε την απόφαση του Σουηδίας ε, να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Θα συζητήσουμε μαζί της λοιπόν για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη λωρίδα της Γάζας. Ε, την επόμενη χρονιά η Σουηδία θα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε όμως μόνο μία χώρα και μια μάλλον μικρή χώρα. Δεν υπάρχει μια γρήγορη λύση προκειμένου να πείσουμε τις συντηρητικές κυβερνήσεις των κρατών μελών ή και δεξιές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν τα βήματα της Σουηδίας. Ε, θα κάνουμε όμως ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και εκεί που δεν το περιμένει κανείς, ορισμένε φορές ανοίγει ένα παράθυρο, μια χαραμάδα και ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Εμείς λοιπόν στην αντιπροσωπεία μας πάντα προσπαθούμε να βρούμε αυτό το άνοιγμα, αυτή την ευκαιρία, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη μας για τη Γάζα, για την Παλαιστίνη. Και πότε πότε κερδίζουμε και κάποιες μάχες και επιτυγχάνουμε μια πραγματική αλλαγή στα όσα συμβαίνουν. Θα ήθελα όμως να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτή είναι η συζήτηση στη χώρα μου. Τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Ντόναλτ Τραμπ θα είναι πλέον ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας αποσχολήσει καθόλου ή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να δυσκολέψει τα επόμενα βήματα ή είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς εσάς και σας υπόσχομαι ότι θα μιλήσω με τη Σουηδή Υπουργό Εξωτερικών ε, για το θέμα της Γάζας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι από κοινού, αν μπορώ να θέσω εγώ το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στην κυρία Μογκερίνη, φυσικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μη χάνετε την ελπίδα σας όμως, αλλά βέβαια όλα αυτά θα χρειαστούν ε, χρόνο. Δυστυχώς για τους Έλληνες, τους Ελληνοκύπριους, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, οι κυβερνήσεις μας δεν έχουν κάνει αυτά τα οποία έχει κάνει η Σουηδία. Μπορούμε, εν περιπτώσει, βέβαια έχουμε μια κάποια πολιτική ελευθερία και μπορούμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας και μπορούμε επίσης να πιέσουμε και τη Μογκερίνη, όπως επίσης είπαμε και στον κύριο Τζεντιλίνη που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, τον ειδικό αντιπρόσωπο, Του είπαμε ότι είναι ιδιαίτερος μετριοπαθής ε, η γραμμή την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έδωσε απαντήσεις, δεν έδωσε σχόλια ε, για τις εξαγωγές προϊόντων σαν παράδειγμα από το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κατεχόμενα. αναφέρθηκε στην κατανομή αρμοδιοτήτων γύρω από τα θέματα αυτά ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κανονισμός ε, για τέτοιου είδους προϊόντα, σαν παράδειγμα στην Γαλλία, έτσι ώστε να υπάρξει σωστή σήμανση και ετικετοθεσία των προϊόντων που προέρχονται από τα κατεχόμενα. Αλλά άλλα κάνει η Γαλλία, άλλα κάνει ή δεν κάνει μια άλλη χώρα. Υπάρχει μια σύγχυση γενικά. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις έτσι ώστε όταν υπάρχουν παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου οι κυρώσεις να είναι αντίστοιχες του ύψους της παραβίασης και τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τις κοινοτικές διατάξεις. Πρέπει λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει. Έγινε ήδη μία πρόταση να στείλουμε μια επιστολή προς τους Υπουργούς και προς το Συμβούλιο. Ξέρουμε επίσης και την πρόταση για τη διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης, της εταιρικής σχέσης μάλλον, να διακοπεί η λειτουργία της Νομίζω ότι το σουηδικό παράδειγμα, αν μη τι άλλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία μορφή πίεσης εις βάρος των υπόλοιπων κυβερνήσεων, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σταματήσει ο αποκλεισμός της Λωρίδας, γιατί δυστυχώς ακούσαμε φρικτές λεπτομέρειες σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς πολύ πια, γι' αυτό παρακαλώ θα σας δώσω το λόγο πάλι στη Γάζα που μας ακούτε πολύ υπομονετικά. Θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια μικρά ή κάποιες απαντήσεις και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην Πατρίσια. Λοιπόν, στη Γάζα έχετε για λίγα λεπτά ξανά το λόγο. Λέγομαι Μοχάμεντ Αλμπακρή, Διευθυντής ε, της Επιτροπής Γεωργίας στη Γάζα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της συνάντησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια. ان المجتمع الدولي قدم الكثير لقطاع غزة من την υποστήριξη προς την ε, ε, Γάζα, ε, η διεθνής κοινότητα έδωσε κονδύλια στην Παλαιστίνη, αλλά δεν αρκούν τα κονδύλια. Πρέπει να σταματήσει ο αποκλεισμό και ο αποκλεισμό δεν είναι ανθρωπιστικό πρόβλημα, είναι πολιτικό πρόβλημα. Αν ε, λάβατε υπόψη ότι θεωρείστε απλώς ανθρωπιστικό πρόβλημα, είναι σαν απλώς να δίνεις φαΐ σε έναν άστεγο. Δεν αρκεί όμως αυτό. η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτή τη λογική της ανθρωπιστικής βοήθειας και μόνον χωρίς ε, να υπάρξει μια σαφής πολιτική τοποθέτηση. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι αυτή η πολιτική τοποθέτηση. Ε, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες προσφέρουν μεν χρήματα αλλά δεν προσφέρουν πολιτική υποστήριξη. Και ε, Πρέπει βέβαια να πούμε ότι η Ευρώπη ναι μεν πρόσφερε πολιτική υποστήριξη αλλά δεν αρκεί. Η Γαλλία έχει μια πολύ θετική ε, στάση την οποία θέτησε, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα αλλά ε, θα θέλαμε πραγματικά και άλλες χώρες ε, να κάνουν αυτό που έκανε η Γαλλία. Να μποϊκοτάρει δηλαδή τα Ισραηλινά προϊόντα τα οποία παράγονται στους ε, περιοχές, στις περιοχές ε, των επικισμών. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις ουσιαστικά μας στερούν ε, τα τρόφιμά μας, διότι κατάσχουν τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις. Για την ερώτηση όσον αφορά τον Ντόναλτ Τραμπ, ειλικρινά εμείς έχουμε κυριευθεί από το φόβο. Έχουμε δει βέβαια την αλληλουχία ε, των Αμερικανών Προέδρων και αν ναι, καθένα οι πολιτικές τους δεν ήταν ε, υπέρ της Πανελληστίνης αλλά υπέρ ε, του Ισραήλ. Ειλικρινά δεν πιστεύουμε ότι θα έρθει λύση από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της ενώπιον της ανάγκης να προστατεύσει τον Παλαιστινιακό λαό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον ε, ε Παλαιστινιακό λαό όταν υπάρχει κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, ε, κατάσχονται οι εκμεταλλεύσεις τους, ε, η επισητιστική κατάσταση είναι φρικτή, η οικονομική κατάσταση επίσης. Η διεθνής κοινότητα, κυρίες και κύριοι, δεν έχει κουνήσει το μικρό της δαχτυλάκι, δεν έχει πιέσει το Ισραήλ και δεν αντιλαμβανόμαστε και για ποιο λόγο. Έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι η λύση θα έρθει μόνο όταν υπάρξει πραγματικά ε, ισχυρή πίεση. Δεν θα μπορέσει να έρθει λύση από το Ισραήλ. Πριν δώσω το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο για να θέσει μια ερώτηση για τη Χαμάς. Καλησπέρα σας. Είμαι υπεύθυνο ε, της Εξωτερικής Υπηρεσίας Δράσης για την ε, Παλαιστίνη. Να σας ευχαριστήσω και για τις παρεμβάσεις σας. Τις εκτιμούμε ιδιαίτερως, αλλά αυτό το οποίο εκτίμησα περισσότερο είναι τα σχόλια και περιγραφές από τους φίλους μας στη Γάζα. Ε, δεν ξέρω πόσες γυναίκες αλληλείς έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εξαιρετικό το γεγονός αυτό. Και πραγματικά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό. Άκουσα πολύ ε, καλά, προσεκτικά την περιγραφή της καθημερινής σας δουλειάς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Και θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε ε, το θέμα της Γάζας ε, πάρα πολύ προσεκτικά. Στις 29 Νοεμβρίου, πολύ πρόσφατα, ο πρέσβης μας, επικεφαλής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, ε, δημοσίευσε μια επιστολή επί τη ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και εκεί υπάρχει μια μακρά παράγραφος ε, την, η οποία ζητά να ανοίξουν οι διάβλοι για αγαθά, πρόσωπα και υπηρεσίες. Ε, επομένως, ε, εμείς και πάλι αναλαμβάνουμε αυτή τη δέσμευση. Σήμερα όμως δεν έχει γίνει συζήτηση για ένα άλλο ακαθόδες ζήτημα και το οποίο δεν θίγει κανείς, που είναι η Χαμάς, που είναι το άλλο ζήτημα το οποίο αφορά τη Γάζα. Λυπάμαι που σας το λέω έτσι, αλλά δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και για το θέμα αυτό. Όσο σημαντική και απαραίτητη είναι η συζήτηση για την ανθρωπιστική βοήθεια, και την οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν θέλω να είμαι αρνητικό ω προ αυτό. Κάθε άλλο. Θέλω να είμαι θετικό ω προ τη συγκεκριμένη πτυχή. Ξέρετε ότι η ΧΑΜΑΣ και πάλι εξακολουθεί να θεωρείται από το Συμβούλιο ω τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχει βέβαια διέξοδο, ίσω όχι τι επόμενε δύο εβδομάδε, αλλά ε, μεσοπρόθεσμα και έχουμε και κάποιες θετικές ενδείξεις ε, από το συνέδριο της ΦΑΤΑΧ. Όχι επισήμως ανοιχτά, αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι η ΦΑΤΑΧ θα ήταν διατεθειμένη να κινηθεί ε, προς ε, μια διαδικασία συζητήσεων με τη Χαμάς για τις μελλοντικέ εξελίξεις εντός της Παλαιστίνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να χάσουμε από αυτή τη συζήτηση ε, και ε, να το περιλάβουμε και αυτό στη συνολική εικόνα όταν συζητάμε το ζήτημα. Ήθελα να το θίξω και αυτό για να είναι πλήρη η συζήτηση και από αυτή τη σκοπιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ε, δεν αναπτύχθηκα αρκετό. Όταν ήμουν στο συνέδριο της Φατάχ, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε ήταν ότι υπήρξε μια δήλωση της Χαμάς, την οποία διάβασε ο επικεφαλής της Χαμάς στο συνέδριο της Φατάχ, ε, και υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει δυνατότητα για εθνική συμφιλίωση μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο βέβαια να συνεργαστούν όλοι και θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος έστειλε ε, δήλωση στο συνέδριο της ΦΑΤΑΧ και ε, διαβάσαμε τη δήλωση αυτή εκεί. θα δώσω πρώτα το λόγο στην Πατρίτσια και μετά ε, επειδή είναι και η Αντζελίνα εδώ, θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Η Πατρίτσια. Ένα λεπτό μόνο. Βρισκόμαστε σε κατεπίγουσα κατάσταση στη Γάζα. Η λωρίδα της Γάζας ε, πλήττεται και είναι ε, πολύ πιο ευάλωτοι η κάτοικοι της Γάζας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δράσουμε όσο υπάρχει ακόμα περιθώριο λιγμών, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει ε, την επόμενη χρονιά ή σε δύο χρόνια. Η πρότασή σας, ε, αν γίνει αποδεχτή από την Πρόεδρο, θα μπορούσε να βοηθήσει. Υπάρχει στο διεθνές δίκαιο μια σειρά διατάξεων που λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα όταν υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, διασφαλίσουν ότι θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Έχω και το σχετικό άρθρο εδώ μπροστά μου. Η κυρία Άντερσον συμφωνεί ε, θα πρέπει να σταλεί μια επιστολή σε όλα τα κράτη-μέλη για να υπενθυμίσουμε τις ευθύνες τους ε, στην παραμονή των 50 ετών ε, της κατοχής ε, ε, πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Ξέρω φυσικά ότι δεν είναι η άποψη αυτών που βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά το μήνυμα το οποίο πρέπει να διαβιβάσουμε είναι ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε τη Γάζα από το στόχο μας, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος αύριο η ασφυξία αυτή, αν συνεχιστεί, η ανθρώπινη και οικονομική ασφυξία, μπορεί αύριο να μην υπάρχει κανένα περιθώριο λιγμών. Η Πατρίσια θα προετοιμάσει την επιστολή και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Συμπερασματικά, μου επιτρέπετε, να πω ότι εγώ πηγαίνω στα κατεχόμενα τα τελευταία 15 χρόνια. Η κατάσταση πάρα πολύ απλά χειροτερεύει. Η πίεση από τους επικισμούς είναι πάρα πολύ ψηλή στη Δυτική Όχθη και τα προβλήματα στη Γάζα τα είδαμε. Η απόγνωση των Παλαιστινίων αυξάνεται και απέναντι στην δική τους πολιτική εξουσία, απέναντι κυρίως στις δυνάμεις κατοχής, αλλά και απέναντι στις ΜΚΟ. Όλο και περισσότερη κριτική απέναντί μας. Εμείς πήγαμε εκεί πριν 10-15 χρόνια για να τους βοηθήσουμε να συνέλθουν υποτίθεται. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι πολύ περιορισμένο. Εμείς στην ουσία είναι σαν να τους δίνουμε λευκοπλάστη για τα τραύματά τους. Τίποτα περισσότερο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόποση και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσία των κρατών μελών βλέπουμε την κόπωση και των ίδιων των Παλαιστινίων δυστυχώς. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη ή στη Λωρίδα. Δυστυχώς μπορούμε να προγραμματίζουμε στην Δυτική Όχθη για κάποιες εβδομάδες, μήνες ή έστω και λίγα χρόνια, αλλά δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε στον Παλαιστινιακό πληθυσμό μια ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης. Είναι προφανές, αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι σχετικά με την Δυτική Όχθη, αλλά κυρίως με τη Γάζα, ας μην περιμένουμε να δράσουμε μετά από πολιτική βούληση και μετά από πολιτική λύση. Η πολιτική λύση θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο. Οι άνθρωποι εκεί καθημερινά υποφέρουν, τώρα υποφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν την αίσθηση αυτής της κόπωσης και οργανώσεις σαν τη δική μας θα συντατικοποιήσουν τη δράση τους έτσι ώστε να βοηθήσουμε έστω και στη μικρή αυτή κλίμακα. Θα ήθελα λοιπόν εξ ονόματος όλων εδώ όλοι εδώ οι βουλευτές, η πλειοψηφία θα έλεγα στην ουσία απευθύνει αισθήματα αλληλεγγύης απέναντί σας, κατανοούμε την κριτική που ασκείται απέναντί μας, αλλά πραγματικά απέναντί σας έχετε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία η οποία δεν θα το βάλει κάτω. Και εμείς νιώθουμε μια απόγνωση μερικές φορές, νιώθουμε ότι δεν κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αλλά η δυσφορία αυτή που νιώθουμε δεν πρέπει να σας εμποδίζει να κατανοήσετε εσείς εκεί στη Λωρίδα ότι υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι που θέλουν να σταματήσει η κατάσταση αυτή και δεν πρέπει το Ισραήλ να συμπεριφέρεται με την ατιμορρησία αυτή η οποία γύρω του δυστυχώς του το επιτρέπει. Πρέπει λοιπόν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να τιμήσουν τις ανηλυμένες τους υποχρεώσεις και το κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί πλήρως. Δυστυχώς, αν δεν αυξήσουμε την πολιτική μας δράση, έστω και με το κεφάλι εμείς θα χτυπήσουμε τον τοίχο που έχουμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Είναι δικαιολογημένη η κριτική την οποία ασκείται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όσους σας βοηθούν. Αλλά ταυτόχρονα να ξέρετε ότι εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση, βλέπουμε τα προβλήματά σας, βλέπουμε τα προβλήματα με τον επικισμό Βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νομαδικές φυλές των Βεδουίνων επίσης και σαν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και οι αντιπρόεδροι θα ήθελα να πω ότι δεν περνάει μία μέρα που να μην κάνουμε κάτι έστω και μικρό για την Παλαιστίνη και δεν περνάει μία εβδομάδα που τα μέλη του Κοινοβουλίου να μην ασχολούνται με την Παλαιστίνη. Δεν το κάνουμε όσο οργανωμένα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι η κοινοβουλευτική μας αντιπροσωπεία θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι δεν θα σας εγκαταλείψουμε. Θα δώσω το λόγο, θα δώσουμε τώρα στην Αντζελίνα να δούμε ένα μικρό βίντεο ενός λεπτού για τους Βεδουίνους. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των κοινοτήτων των Βεδουίνων στο Στρασβούργο επαναλαμβάνω Θέλουμε να κατανοήσουμε όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν ανοιχτά στην περιοχή σας και να είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να κοπεί η σύνδεση με τη λωρίδα της Γάζα. θα προσπαθήσουμε να έρθουμε στη Γάζα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, δεν μας επιτρέπουν προς το παρόν αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Τον Φλεβάρι εμείς θα δοκιμάσουμε πάλι και η δική μου πολιτική ομάδα έτσι ώστε του χρόνου όλες οι πολιτικές ομάδες και όλες οι αντιπροσωπείες που έχουν κάποια σχέση με τη Λωρίδα να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση. Και η τεχνολογία ευτυχώς λειτουργεί εις βάρος των άλλων. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες σας και για την μοναδική γυναίκα που ψαρεύει που έχω γνωρίσει εγώ τουλάχιστον να συνεχίσει την προσπάθεια και να προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο.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 δώσουμε το λόγο σε εσά και σας ευχαριστούμε που μας δώσετε τη δυνατότητα να το δούμε. Ε, κανονικά θα ήμουν εδώ με δύο Βεδουίνους συναδέλφου. Δυστυχώ ακόμα δεν έχουν ε, δοθεί οι θεωρήσεις διαβατηρίων τους. Ε, μάλλον θα τις λάβουν αυτή την εβδομάδα, αλλά θα διαβάσω τη δήλωσή τους. Αυτή είναι η δήλωση που θα είχαν κάνει ο Σλεμάν και Τάρικ Κορσάν αν ήταν εδώ για να μιλήσουν για τα δικαιώματα των Βεδουίνων στη Δυτική Όχθη. Όπως γνωρίζετε, οι Ισραηλινές αρχές έχουν εκδώσει ε, εντολές κατεδάφιση σε περισσότερες από τις κοινότητές μας, ιδίως σε ανθρωπιστικές δομές τις οποίες έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που κόστησαν εκατομμύρια ευρώ. Ε, κατεδάφισαν ολόκληρες κοινότητες. Για παράδειγμα, 8 κατοικίες οι οποίες ανήκαν στην οικογένειά μας ε, τον Οκτώβριο και δεν επιτρέψουν και στους Βεδουίνους να κτίσουν τίποτα ή να επισκευάσουν σπίτια ε, τα οποία είναι φτιαγμένα από κασίτερο και ε, χαρτί, χαρτόνι. Ε, τα παραδοσιακά μας σπίτια καταστρέφονται παραδοσιακά και, τα, και οι άνθρωποι και τα ζώα μένουν έξω στο κρύο, πεθαίνουν τα ζώα και αυξάνεται η θάνατος και οι ασθένειες μεταξύ των λαών μας. 11.000 εντολές κατεδάφισης ε, κρεμούν ε, στα σπίτια, τα σχολεία μας και στα ε, καταφύγια για τα ζώα στην ζώνη Γ. Τα στατιστικά στοιχεία χειροτερεύουν κάθε μήνα ε, καταδοφίζονται συγκεκριμένε δομέ, οι οποίε έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτο είχαμε τι περισσότερε καταδαφίσει από το 2009, αύξηση τη τάξη του 63% από το 2015. Από 1η Ιανουαρίου του 2016, 1.054 δομέ καταδαφίστηκαν, εκτοπίστηκαν 1.598 άτομα και επηρεάστηκαν 6.436 άτομα. Φέτος περίπου 30% των δομών που καταδαφίστηκαν, ε, έχουν χρηματοδοτηθεί από χορηγούς και 33% ήταν βεδοίνων. Τον ε, Ιούλιο σε μια διάσκεψη ε, της Κνεσέτ για τη ζώνη ΓΑΜΑ... ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι είναι αντίθετο με τις συμβάσεις της Γενέβης, τις ειρηνευτικές διαδικασίες του Όσλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αποκάλεσε ε, ένας καθηγητής ε, του Ισοξφόρδης, η Ντόουν Τσάτι, ε, πολιτιστική γενοκτονία. Ο πρόεδρος ε, Αραφάτ αναφέρθηκε στους Βεδουίνους ως ε, τους θεματοφύλακες του Ιερουσαλήμ και, της Ιερουσαλήμ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι είναι ήδη ασταθή η Μέση Ανατολή. Το να σταματήσουμε λοιπόν τα ευρύτερα σχέδια της Ιερουσαλήμ ε, για το ε1 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εμείς οι Βεδουίνοι είμαστε πράγματι οι φύλακες μιας βιώσιμης Παλαιστίνης. Οι αρχές κατοχής ε, σκοπεύουν να εκτοπίσουν Βεδουίνους στον ΟΕΜΕΝ δίπλα σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής ε, και είναι η μεγαλύτερη διαδικασία εκτοπισμού. Αναφέρονται ελεύθερα στην προσάρτηση της ζώνης Γ, που είναι το σύστημα στήριξης για τις ζώνες Α και Β. Εμείς ως Βεδουίνοι φυσικά απορρίπτουμε αυτά τα σχέδια, μας πλήττουν φρικτές οικονομικές συνθήκες, έλλειψη πρόσβασης σε βοσκοτόπους, σε ίδρυυση, ε, λόγω της επέκτασης των επικισμών και των μικρών κλειστών στρατιωτικών ζωνών που εκτείνονται σε όλη την περιοχή. Ε, υπάρχει και ένα φράχτης διαχωρισμού και δεν μας επιτρέπει πρόσβαση στην Ιερουσαλήμ που ήταν η βασική μας αγορά για να πουλούμε τα προϊόντα μας. Ε, δεν έχουμε υποδομές, ηλεκτροδότηση, τρεχούμενο νερό, δεν υπάρχει πρόσβαση στα οδικά δίκτυα και προβλήματα για τα παιδιά μας, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο ή σε ιατρικά κέντρα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ένδυα και ανεργίας και πολύ χαμηλό ποσοστό παιδεία. Ζητούμε λοιπόν πραγματικά να πιέσετε το Ισραήλ να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις των κοινοτήτων μας, ε, των καταφυγίων για τα ζώα μα, τα σπίτια μα και τα σχολεία μα. Ζητάμε να προσφέρετε πραγματική προστασία για να σταματήσουν τα σχέδια εκτοπισμού και επίσης ζητάμε βασικές υπηρεσίε: παιδεία, κατάλληλη στέγαση και υγειονομική περίθαλψη, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας ελεύθερα, χωρίς το συνεχή φόβο και την ανασφάλεια. Ευχαριστώ, παρακαλώ βοηθήστε μα. Κυρία Πρόεδρε, η δική μου δήλωση ε, σε απάντηση στην ερώτησή σας, τι μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι εγώ ως ε, ακτιβίστρια για την ειρήνη ε, στο Ισραήλ και ως ακτιβίστρια τα τελευταία 25 χρόνια θα ήθελα να πω το εξή: Χωρίς πραγματική διεθνή πίεση χειροτερεύει η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλη βία και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ε, κυρίως οι πολιτικές κατεδαφίσεων που είναι τμήμα της επέκτασης που προωθούμε δημιουργούν ένα κλίμα στο οποίο οργιάζει η τρομοκρατία και ε, από πλευράς Ισλαμικού κράτους. Η παρουσία μου εδώ σήμερα που μιλώ κατά της κατοχής των 50 ετών που ε, θέτει σε κίνδυνο τα δημοκρατικά συμφέροντα του Ισραήλ και τις εβραϊκές αξίες. Είναι κάτι ε, το οποίο θα ποινικοποιήσει το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και η κοινωνία των πολιτών σιωπά. Δηλώσεις ή απειλές έχουν αποδειχθεί ανίκανες να αλλάξουν τις πολιτικές του Ισραήλ και από τους επικιστές, ε, οι οποίοι ε, στο 15% τους είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θεωρούνται ως καλές δράσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν να υπάρξει λογιδοσία και ε, πράξεις, διότι τα λόγια δεν οδηγούν σε τίποτα δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν ανίποτες πολιτικές του Ισραήλ που δεν σταμάτησαν τις, τους εκτοπισμούς των Βεδουίνων στη ζώνη Α. Περιμένουμε ότι θα κλιμακωθούν οι εκτοπισμοί αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από πλευράς Ντόναλτ Τραμπ. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι η νομιμοποίηση ε, των επικισμών μπορεί να οδηγήσει στη Χάγη. Και την προηγούμενη εβδομάδα, ε, σε ένα φόρουμ το οποίο έγινε, αναφέρθηκε ε, η νομιμοποίηση αυτών των περιοχών. Όλο αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πιθανή ποινικοποίηση αλλά ε, οι κυβερνητικοί ε, οι οποίοι έχουν μονή με την εξουσία εξακολουθούν να προχωρούν ακάθεκτοι. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι περισσότερο σημαντικό για λογοδοσία ε, όσο εκτοπισμός αθών πολιτών. Παρεπιπτόντων, στο 60% των ανθρώπων στη Γάζα ήταν ευεδοίνοι πρόσφυγες οι οποίοι διέφυγαν. Αυτό το θέμα του εκτοπισμού των Βεδουίνων είναι έγκλημα πολέμου, είναι και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ε, πραγματικά ε, συμμετέχουμε σε αυτά τα εγκλήματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα σταματήσουμε ακόμα και πιστεύω ότι όλοι εσείς έχετε τη δύναμη και την εγγενή δέσμευση προς την ανθρωπιά λόγω της συμμετοχής σας σε αυτή την αντιπροσωπεία να υποστηρίξετε αυτές τις παγκόσμιες αξίες, ε, τις οποίες ίσως αυτή τη στιγμή μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε κλήσεις για αποζημίωση που έρχονταν από την ομάδα εργασίας ε, του Ομπάμα, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πολιτικές. Να χρησιμοποιηθεί το θέμα της ευθύνης των τρίτων χωρών και η εφαρμογή της δικής σας της νομοθεσίας. Να εφαρμόσετε την ειδική έκθεση που κάνουν επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο για την περιοχή της Γάζας και τη ζώνη Γάμα. Δεν εφαρμόζονται όλα αυτά και από ό,τι καταλαβαίνω λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Οι διπλωμάτε επιτόπου λοιπόν εδώ και 10 χρόνια ζητούν πράγματα τα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν. Και για να σα παραθέσω το, κάτι του Τζον Fitzgerald Kennedy, αν δεν το κάνουμε εμεί, ποιοι, αν δεν το κάνουμε τώρα πότε. Ερωτήματα τα οποία παρεπιπτόντω ξεκίνησαν τη δική μου την πορεία ω ακτιβίστρια στο Σιναή στην Αίγυπτο με του Βεδουίνου πριν από 25 χρόνια. Και τέλο, θα ήθελα να ε, μιλήσω για τους λεγόμενους φίλους του Ισραήλ που μπορεί να βλέπουν από ε, κάμερα μέσω διαδικτύου. Οποιοςδήποτε φίλος του Ισραήλ θα πρέπει να πει στην Ισραηλινή κυβέρνηση ότι και οι στενότεροι σύμμαχοι δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν ε, ε, και να μην φτάσει το θέμα αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε συναντήσεις, ε, διαζώσεις μαζί σας, ελπίζοντας και να έχουμε και την παρουσία των Βεδουίνων φίλων μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. που διαβάσατε και τη δήλωση εξ ονόματος των Βεδουίνων φίλων που δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι ανάμεσά μας εδώ. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καταλαβαίνουμε επίσης και την προσπάθεια που κάνετε εσείς. Ζητάτε για μεγαλύτερη πίεση, ζητάτε για μεγαλύτερη προστασία, δεν ζητάτε πολλά και όμως για τους Βεδουίνους όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, η κατάσταση είναι πολύ κακή. Σε ένα από τα τελευταία ταξίδια μας εκεί, είδαμε επίσης ε, τις επιπτώσεις ε, των δράσεων των ε, επίκων στην περιοχή, εις βάρος των Βένων, μου είπαν οι Βεδουίνοι ότι αν οι γίδες τους περάσουν από τη μία πλευρά του χωματόδρομου στην άλλη και πάνε να φάνε χόρτο από την απέναντι, συλλαμβάνονται οι γίδες, φυλακίζονται οι γίδες και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της γίδας να πληρώσει για την απελευθέρωσή της. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως έχει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την τεράστια προσπάθεια και στήριξη που δίδεται στους πληθυσμούς αυτούς Ο κύριος Μαρτά ε, είχε φέρει στο Στρασβούργο κάποιους από την κοινότητα των Βεδουίνων. Ευχαριστώ Μαρτίνα. Είχαμε υποδεχθεί τον κύριο Αμπουσάκ. Ο Αμπουσάκ μας είπε πώς έχει η κατάσταση σήμερα, ποια είναι η πραγματικότητα για τους Βεδουίνους και για την απαγόρευση πρόσβαση σε υδάτινους πόρους των Παλαιστινίων και των Βεδουίνων. Ε, για την παρατήρηση που κάνατε, δεν θέλω να έρθω σε αντίθεση μαζί σας, αλλά θα έλεγα ότι σε σχέση με τους Βεδουίνους γίνεται η προσπάθεια να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τους Γκαζαουί. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι φοβάμαι μάλλον ότι αν θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία, δεν ξέρω αν όσο ζούμε θα τη δούμε, είναι σαφές ότι θα πρέπει πλέον να χτυπήσουμε όλες τις πόρτες, να δούμε αν εμείς σαν πολίτες, ούτε καν σαν βουλευτές, σαν πολίτες, να δούμε τους υπουργούς δικαιοσύνης, διότι εδώ υπάρχει έλλειψη συνδρομής σε ε, άνθρωπο σε κίνδυνο, σε ανθρώπου σε κίνδυνο. Θα πρέπει οι Βεδουίνοι να ξέρουν ότι τους στηρίζουμε. Η Μαρτίνα εδώ και χρόνια πηγαίνει εκεί και περνάει ώρες ολόκληρες παρεμποδιζόμενοι και ελεγχόμενοι στους αερονημένες τους Ισραηλινούς. Αλλά δεν έχει σημασία, αναζητούμε πάντα λύσεις στους λαούς που υποφέρουν. Και στρέφομαι εδώ και στον ίδιο μου τον εαυτό. Αυτό το κοινοβούλιο, αυτό το όργανο, ακόμα και αν δεν έχει αποφασιστική άποψη ε, θα έλεγα μέχρι τώρα, νομίζω ότι σιωπά εμπολής και η πρόταση την οποία θα κάνουμε ελπίζω να γίνει δεκτή. Δεν θα υπογραφεί μόνο από αυτήν εδώ την αντιπροσωπεία, θα πρέπει να την προτείνουμε προς ψηφοφορία στους 751 βουλευτές, έτσι ώστε κάθε Ευρωπαίος πολίτης, ανεξαρτήτως της άποψης που έχει για την Παλαιστίνη και τη Γάζα, να γνωρίζει το τι υποστηρίζει ο βουλευτής του. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο σκύλος γαυγίζει, το καραβάνι περνάει, φοβάμαι ότι πολλά καραβάνια έχουν περάσει και δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Ο κύριος Πρέσβης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Στη συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Μαρτά. Όταν βλέπει κανείς την κατάσταση στην Παλαιστίνη, εγώ παρακολουθώ άλλωστε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και 16 χρόνια. Έχω δει το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Παλαιστίνη. 50-49 χρόνια κατοχής έχουμε βιώσει. Και αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι αν κάποιος αυτήν εδώ την αίθουσα δεν συμφωνεί μαζί μου να μου το πει, γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ και 49 χρόνια είναι η στρατιωτική κατοχή. Αυτή είναι η πρώτη σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Εδώ και δύο εβδομάδες άκουσα τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών που είχε πάει στη Γάζα. Τρεις φορές είπε ότι η Γάζα είναι ένα γκέτο. Εδώ υπάρχει δηλαδή έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Διεθνές Ποινικό. Αν διαφωνείτε να μου το πείτε. Εγκλήματα πολέμου διαπράττει το Ισραήλ κυρίες και κύριοι εδώ και 49 χρόνια. Οι επικισμοί, η κατάσταση ε, των Βεδουίνων όπως είπε η Άντζελα. Εγκλήματα πολέμου, μαζικά εγκλήματα πολέμου εδώ και 49 χρόνια. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει γενοκτονία ή κάτι άλλο. Για τους Βεδουίνους ναι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι έγκλημα εις βάρος της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι η συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ εδώ και 49 χρόνια. Διερωτώ λοιπόν για την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ξέρουμε τι κάνει το Ισραήλ εδώ και 49 χρόνια, αλλά αυτό που λέω εγώ εδώ το 2000 και μετά είναι ότι οι οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και το Ισραήλ ενισχύονται. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, ξέρουμε ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι η συμπορά του Ισραήλ, αλλά πρέπει να του πούμε αυτό. Γιατί τι κάνει η διεθνής κοινότητα, πώς συμπεριφέρεται η διεθνής κοινότητα. Αυτή η παθητική αντιμετώπιση δυστυχώς ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει σε τέτοιου είδους εγκλήματα. αν δεν επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί το Ισραήλ να αλλάξει άποψη. Δυστυχώς σήμερα η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παθητική, αλλά νομίζω ότι και έμεσα ενθαρρύνεται το Ισραήλ. Εγώ παρακολούθησα τις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Μπορείτε να μου πείτε σήμερα γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν συμμετέχουν έτσι ώστε να ζητήσουν να διαγραφεί το σημείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί δεν συμμετέχει στη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν συμμετέχει όταν ψηφίζουμε την έκθεση της ε, Επιτροπής Έρευνας για τη Γάζα. Οι χώρες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης σιωπούν Αυτά ενθαρρύνουν τη συνέχιση της εγκληματικής συμπεριφοράς του Ισραήλ. Δεύτερον, και θα ήθελα ίσως να ξεκινήσω από αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνετε, για τη στήριξή σας και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δυστυχώς όμως αν δεν φανούμε αυστηροί απέναντι στο Ισραήλ δεν θα αλλάξει στάση το Ισραήλ και θα συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάσταση εις βάρος της Παλαιστίνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ουδέτερος ενώπιον αυτής της κατάστασης και φυσικά η απραξία δεν είναι ε, επιλογή. Εμείς λοιπόν σε αυτή την αντιπροσωπεία ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα συνεχώς να επιταχύνει τις διαδικασίες της και πιστεύω πραγματικά ότι τα κράτη-μέλη που ε, εστάλησαν εδώ, οι ευρωβουλευτές που εξελέγησαν, ήρθαν για κάποιο λόγο. Επειδή υπάρχει ε, συνήθως λίστα ε, σε κάποια κράτη-μέλη, δεν είναι όλοι γνωστοί οι ευρωβουλευτές σε κάποια κράτη-μέλη για αυτό που είναι. Το να βρούμε λοιπόν τη συμπεριφορά τους δεν είναι πάντα ε, κάτι που γνωρίζουν οι άνθρωποι που τους ψηφίζουν και τους στέλνουν εδώ. Πιστεύω ότι οι ευρωβουλευτές ε, θα πρέπει να πιέζονται περισσότερο από τους ε, ψηφοφόρους τους και αν συνέβαινε αυτό θα συμπεριφέρονταν διαφορετικά. Ό,τι είπατε για το Ισραήλ, για τη διεθνή κοινότητα, για το γεγονός ότι δεν γίνονται αρκετά. Υπάρχουν κάποια ψήγματα ελπίδας, άμα δούμε τι συνέβη στη Σουηδία, τουλάχιστον να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη. Ε, αν καταφέρουμε να τον αναγνωρίσουν όλα τα κρατημέλη, αν καταφέρουμε το Ισραήλ ε, να είναι υπόλογο για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ε, αν η διεθνής κοινότητα κάνει πολύ περισσότερα, πολύ πολύ περισσότερα, τότε αντί λοιπόν να ενθαρρύνουμε και όντως να είμαστε και σχεδόν συνένοχοι για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι και εμείς είμαστε υπεύθυνοι εξίσου γιατί δεν κάνουμε αρκετά. Και το φωνάξαμε, χτυπήσαμε τη γροθιά μας, υψώσαμε τη φωνή μας, ε, λάβαμε δράσεις, λάβαμε μέτρα και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετοί ευρωβουλευτές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να κάνουν αυτό που είναι σωστό, αυτό που πρέπει. Και νομίζω ότι πρέπει να τους εκθέσουμε στους ψηφοφόρους τους, διότι αν δείτε ε, την αντίδραση στην τελευταία επίθεση στη Γάζα, οποιοδήποτε είχε έστω καρδιά, έστω ανθρωπιά, ε, βγήκε στους δρόμους και διαδήλωσε, διότι ήταν ο μόνος τρόπος που ήξεραν να αντιδράσουν. Ε, αυτό το οποίο λένε όλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα και το τι πρέπει να κάνουν πολύ πολύ περισσότερα, έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην ε, ε, συμμετοχική δημοκρατία και στην ισχύ των ε, ανθρώπων και αν οι πολίτες γνώριζαν τι κάνουν κάποιοι από τους ευρωβουλευτές τους, τότε πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να συμπεριφέρονταν λίγο διαφορετικά και θα ήξεραν και τι να κάνουν, διότι εμάς μας πιέζουν για την DTIP, για τη ΣΥΤΑ, για τα φυτοφάρμακα, για τη νομοθεσία, για οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε επιτροπή και αν εμάς ως ευρωβουλευτές μας πιέσουν οι ψηφοφόροι μας, τότε συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Ε, προσέχουμε πώς ψηφίζουμε όταν φτάνουμε στην Ολομέλεια. Ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι μας ζητούν να ψηφίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δεν συμβαίνει και ε, κατά την άποψή μου αρκετά όσον αφορά την Παλαιστίνη και αυτά τα οποία έχουμε επιτρέψει το Ισραήλ να κάνει και εμείς μπορούμε απλώς να δεσμευθούμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάνουμε εδώ σε αυτή την αντιπροσωπεία. Όλοι είμαστε από διάφορες πολιτικές ομάδες, έχουμε διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό παρελθόν και διαφορετικές πεπιθήσεις και πραγματικότητα, αλλά είμαστε ένα ενωμένο μέτωπο όταν συζητούμε την Παλαιστίνη. Θέλουμε όλοι να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα και θέλουμε η διεθνής κοινότητα όχι μόνο να προσέξει, αλλά να αντιδράσει και να διασφαλίσει ότι ε, το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Ε, ευχαριστώ λοιπόν για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, για την ε, Άντζελα επίσης που έθιξε το θέμα των ε, Βεδουίνων και το βίντεο τους ανθρώπους ε, από τη Γάζα, την οργάνωσή σας. Ε, πραγματικά ε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για σας. Ήσασταν εκεί εδώ και 15 χρόνια γιατί θέλετε να κάνετε περισσότερα, θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα επί επιστόπου και το ίδιο θέλουμε και εμείς. συλλογικά λοιπόν να συνεχίσουμε όλοι να συνεργαζόμαστε, κάτι θα καταφέρουμε. Θέλω να επαναλάβω για τους ευρωβουλευτές που δεν ήταν εδώ πριν ότι θα πρέπει να ενημερώσουν στη γραμματεία μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, αν θέλουν να πάνε στην αποστολή, ε, το ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ορισμένες φορές η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περιορίζει λίγο το έδειργο των αντιπροσωπιών, διότι θεωρούν ότι ε, είναι δικό τους πεδίο ευθύνης. Ε, ορισμένες φορές μας λένε τι ώρες μπορούμε να συνεδριάσουμε και δεν είναι πάντα η καλύτερη στιγμή για όλους τους ευρωβουλευτές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ευρωβουλευτές όμως, γιατί φροντίζουν τουλάχιστον να στείλουν το προσωπικό από τα γραφεία τους όταν δεν μπορούν να παρευρεθούν και ξέρουμε ότι το προσωπικό κάνει πάρα πολλή δουλειά. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς, γιατί δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ε, συνομιλείς χωρίς εσάς. Ε, μείνετε και λίγο χρόνο περιττέρου και σας ευχαριστούμε λοιπόν για το χρόνο που μας προσφέρετε, όχι κάθε βράδυ, αλλά κάθε φορά που έχουμε τέτοιες συνεδριάσεις. Μας δίνετε πολύ γενναιόδωρα κάποια λεπτά επιπλέον. Σας ευχαριστώ πολύ.